Now the first vote is a roll call vote. Η πρώτη ψηφοφορία θα γίνει με ονομαστική κλίση, γι' αυτό παρακαλώ τοποθετήστε τις κάρτες σας στο μηχάνημα. The voting begins. Η μερίσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία σύμφωνα με την απλοποιημένη διαδικασία επί της έκθεσης της αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Επιτροπή Συνδιαλλαγής σχετικά με τον κοινό κανονιστικό πλαίσιο για δίκτυα και υπηρεσίες ηλεκτρονικών επικοινωνιών. Έκθεση Τράουτμαν. Τη θέτω σε ψηφοφορία με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Έχετε ακόμα 10 δευτερόλεπτα για να ψηφίσετε. 10 seconds. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Λήξη ψηφοφορία. Εγκρίνεται με 510 ψήφου υπέρ. Συγχαρητήρια στην κυρία Τράουτμαν. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία επί της έκθεσης ΣΤΕΣ e σύμφωνα με την απλοποιημένη διαδικασία ε, της Αντιπροσωπείας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην Επιτροπή Συνεδριαγής σχετικά με τις στατιστικές για τα φυτοφάρμακα. Με ονομαστική κλίση ο εισηγητής, ο κύριος Στές, e έχει ζητήσει το λόγο. Κύριε Στές, e για δύο λεπτά. Ε, ε, ε, Θα ήθελα να σας ενημερώσω αγαπητοί συνάδελφοι για τη χρήση των φυτοφαρμάκων γιατί στις αρχές του έτους υιοθετήσαμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ένα κανονισμό για την εμπορία των φυτοφαρμάκων. Και έχουμε και μια οδηγία για την ε, βιώσιμη χρήση των φυτοφαρμάκων από την περασμένη κοινοβουλευτική θητεία. Ο κανονισμό αυτό που αφορά τα στατιστικά στοιχεία για, τον, ε, για τα φυτοφάρμακα αποτελεί το την τρίτη πτυχή, το τρίτο σκέλος αυτού του τριπτύχου. Στην προηγούμενη κοινοβουλευτική θητεία υπήρξε ένα πρόβλημα, υπήρχαν πολλές απουσίες και στην ε, δεύτερη ανάγνωση είχαμε ελάχιστους παρόντες, δεν συγκεντρώσαμε απαρτία για να διεκπαιρεώσουμε το θέμα στη δεύτερη ανάγνωση. Και λαμβάνω το λόγο σήμερα, γιατί θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Σουηδική Προεδρία και την Τσεχική Προεδρία, γιατί χάρη στις προσπάθειές τους κρατήσαμε αγαστή συνεργασία μεταξύ Προεδρίας και Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και μάλιστα είχαμε στείλει έκκληση προς την Προεδρία και στους ηγέτες των κομμάτων για να σώσουμε την έκθεση και να επανέλθουμε σήμερα στην Ολομέλεια μετά την Επιτροπή Συνδιαλλαγής. Ευχαριστώ θερμά. Ε, θέτω την έκθεση ψηφοφορία ε, με ονομασία κλίση άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται με 581 ψήφου υπέρ. Συγχαρητήρια στον κύριο Στάση. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει τη ψηφοφορία επί της έκθεση τη κυρίας Γκέριγκερ σχετικά με τον καθορισμό των γενικών κανόνων για τη χορήγηση κοινοτική ενίσχυσης στον τομέα των διευρωπαϊκών δικτύων. Με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία. Εγκρίνεται με 584 ψήφους υπέρ. Συγχαρητήρια στην κυρία Γκέρινγκερ. Η κυρία Μπέρες ζητάει το λόγο. Α, seine Maschine nicht funktionen. Nein? Δεν λειτουργεί το μηχανημά Άρα. Okay. It's, it's, it's recorded in the minutes. Mrs. Beres, you have the floor. Καταγράφηκε στα πρακτικά, κυρία Μπέρες. Το ίδιο πρόβλημα έχω και εγώ, το μηχάνημά μου δεν λειτουργεί. Κύριε Σέβεριν, έχετε ε, τον, λόγο. Θα στείλουμε κάποιον να, φτιάξει το δικό σας μηχάνημα. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει φοφορία σύμφωνα με την απλοποιημένη διαδικασία επί της του κυρίου Κίρκοπ σχετικά με την έκδοση των κανόνων περί εμπιστευτικότητας των πληροφοριών της Europol. Τώρα, Αγαπητοί συνάδελφοι, η Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνη και Εσωτερικών Υποθέσεων προτείνει την απόρριψη της πρότασης απόφασης εάν συμφωνείτε με τη θέση της αρμόδιας επιτροπής πρέπει να ψηφίσετε κατά σαφές if you agree with the position of the civil liberties committee you must vote against it may not sound reasonable but it is μπορεί να φαίνεται παράλογο αν συμφωνείτε να ψηφίσετε κατά αλλά έτσι πρέπει να γίνει Έρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Το Συμβούλιο δεν είναι παρόν, επομένως η έκθεση αναπέμπεται αυτομάτως στην αρμόδια επιτροπή. Έκθεση Intveld σχετικά με τη θέσπιση κανόνων εφαρμογής που διέπουν τις σχέσεις της Europol με τους εταίρους της. Και για αυτήν την έκθεση ισχύει η ίδια διαδικασία. Εάν συμφωνείτε με την απόρριψη πρέπει να ψηφίσετε κατά. Με ηλεκτρονική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται και η έκθεση αναπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή. Έκθεση Albrecht σχετικά με τον καθορισμό του καταλόγου τρίτων κρατών και οργανισμών με τους οποίους η Europol συνάπτει συμφωνίες, ίδια διαδικασία, με ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται και αναπέμπεται στην αρμόδια επιτροπή. Έκθεση του κυρίου Δίας Δεμέρα σχετικά με την έκδοση εκτελεστικών κανόνων για τα αρχεία δεδομένων εργασίας προς ανάλυση της Europol ίδια διαδικασία με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται και αναπέμπτεται στην Επιτροπή. Έκθεση Κέρκοπ σχετικά με τη διαπίστευση των εργασιών εργαστηρίου ανακριτικής. την ε, ε, με συγχωρείτε, μισό λεπτό. η ίδια διαδικασία, αλλά όχι ακόμα για τον κύριο Κίρκοπ, αλλά για την έκθεση Αλφάνο, σχετικά με τη δημιουργία Ευρωπαϊκού Δικτύου Πρόληψης του Εγκλήματος. Με ονομασική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. απορρίπτεται και αναπέμπτεται στην Επιτροπή. Τώρα η έκθεση Κίρκοπ σχετικά με τη διαπίστευση εργασιών εργαστηρίου ανακριτικής. Ίδια διαδικασία με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται και αναπέμπεται στην Επιτροπή. Η μερίσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία της έκθεσης Μορέιρα σχετικά με τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στην Γεωργία. Με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας εγκρίνεται με 550 ψήφους συγχαρητήρια στον κύριο Μορέιρα. Έκθεση Μορέιρα επίσης... Α, με συγχωρείτε. Ε, η κυρία ε, Κόρλισεν ε, ζήτησε τον λόγο. Παρακαλώ. Παρακαλώ, στείλτε μου ένα τεχνικό και το δικό μηχάνημα θα λειτουργεί. Φυσικά, αμέσω θα σα στείλουμε κάποιον. Το ίδιο πρόβλημα έχω και εγώ, κύριε, κύριε Πρόεδρε. Η συσκευή μου δεν λειτουργεί. Το μηχάνημά του τώρα. Ωραία, μόνο τα δύο έχουμε. Λοιπόν, έκθεση Μορέιρα σχετικά με τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στην Αρμενία. Με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 580 ψήφους. Έκθεση Ράνστορφ σχετικά με τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτικής συνδρομής στην Σερβία. Με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται με 583 ψήφου συγχαρητήρια στον κύριο Ράνστορφ. Έκθεση Βίνκλερ σχετικά με τη χορήγηση μακροοικονομικής χρηματοδοτική συνδρομή στη Βοσνία Ερζεγοβίνη με ονομαστική κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται με 583 ψήφου συγχαρητήρια στον κύριο Βίνκλερ. Έκθεση Μπούλμαν σχετικά με το κοινό σύστημα φόρου προστιθέμενης αξίας με ονομαστική κλίση άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται με 596 ψήφους. Συγχαρητήρια στον κύριο Μπούλμαν. Έκθεση Ρόσπακ σχετικά με τη Σύμβαση για την Προστασία του Θαλάσσιου Περιβάλλοντος του Βορειοανατολικού Ατλαντικού Σύμβαση ΟΣΠΑΡ με έχει κλίση άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται με 624 ψήφους συγχαρητήρια στον κύριο Ρόσπαχ. Στην κυρία Ρόσπαχ, με συγχωρείτε. Έκθεση της κυρίας Γκέριγκερ σχετικά με τη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Βασιλείου Δανίας περί επιδόσεως και κοινοποιήσεως δικαστικών και εξοδίκων πράξεων σε αστικέ ή εμπορικέ υποθέσει. Με ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας, ψηφοφορία εγκρινεται με 651 ψήφους. Έκθεση Γκέριγκεν σχετικά με τη συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Κοινότητας και Βασιλείου Δανία για τη διεθνή δικαιοδοσία, την αναγνώριση και την εκτέλεση αποφάσεων σε αστικέ και εμπορικές υποθέσει με ονομαστική κλίση Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 698 ψήφους. Συγχαρητήρια στην κυρία Γκέριγκερ. Έκθεση Φράγα Εστέβες σχετικά με τη θέσπιση σχεδίου ανασύστασης του Χάλιμπα της Γρυλανδίας. Με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται με 638 ψήφους. Συγκαρητήρια στην κυρία Φράγκα. Έκθεση Κότς σχετικά με τη Σύμβαση περί των Διεθνών Σιδηροδρομικών Μεταφορών, Κοτίφθα. Με ονομαστική κλίση, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 640 ψήφους. Συγκαρητήρια στον κύριο Κότς. Έκθεση της κυρίας Βόλης σχετικά με το εφαρμοστέο δίκαιο στις υποχρεώσεις διατροφής με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 617 ψήφους. Συγχαρητήρια στην κυρία Βόλης. Η κυρία Ράπτη έχει το λόγο. Το μηχάνημά σας. Θα στείλουμε κάποιον Χριστό. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία επί της έκθεσης του κυρίου Σβιέφκα σχετικά με την αίτηση υπεράσπισης της ασυλίας και των προνομίων που υπέβαλε ο Τομπάιας Φλούγκερ, ο οποίος δεν είναι πλέον μέλος. Δεν ξέρω αν η αρμόδια επιτροπή επιθυμεί την απόσυρση αυτής της έκθεσης. Όχι. Εν τη περιπτώσει ψηφίζουμε της έκθεσης, τη θέτω σε ψηφοφορία με μοναδική κλίση ποιοι είναι υπέρ, ποιοι είναι κατά, αποχές, εγκρίνεται. Η μερίδια διάταξη προβλέπει ψηφοφορία επί του κυρίου Σέιερ σχετικά με την προσαρμογή στην κανονιστική διαδικασία με έλεγχο μέρος πέμπτο. Θα ήθελα να σας επισημάνω ότι οι τροπολογίες 1 έως 10 έχουν αποσυρθεί. Οπότε θέτουμε σε ψηφοφορία την πρόταση ως μη αναθεωρημένη. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές απορρίπτεται. Ζητάμε την Επιτροπή αν ε, θέλει κατόπιν αυτού να αποσυρθεί η πρότασή της. Θέλει ο κύριος Ζέιερ το λόγο. Ο κύριος... Ναι. Κύριε Δήμα. I think that we shall not uh, withdraw the proposal. Νομίζω ότι δεν θα πρέπει να αποσυρθεί η πρόταση. Ευχαριστώ πολύ. Επομένως τώρα συνεχίζουμε στις ε, ψηφοφορίες ε, ε, τροπολογιών 11 και 12 που ακολουθούν. Τροπολογία 11 στην παράγραφο 2. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Μετά την παράγραφο 2 ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. Και η τελική ψήφος με ονομαστική κλίση. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 622 ψήφους υπέρ. Τέλος. Η ημερήσια διάταξη προβλέπει την ψηφοφορία της έκθεσης του κυρίου Άλβαρο σχετικά με την χρήση της πληροφορικής στον τελωνιακό τομέα. Ο κύριος Λούχαν έχει ζητήσει το λόγο πριν την ψηφοφορία στην έκθεση. Κύριε Λούχαν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε από πλευρά του ΕΛΚ θα ήθελα να ψηφίσουμε χωριστά την τροπολογία 27. Αφορά την πλήρη πρόσβαση στη Eurojust και στη Euroball στη βάση δεδομένων. Και ήθελα όλοι οι συνάδελφοι να καταψηφίσουν αυτό το σημείο, αυτή την τροπολογία. Έχετε ξεπεράσει δυστυχώς ε, την ε, καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση τέτοιου είδους αιτήσεων. I see you understand Greek very well apparently. Έχετε ξεπεράσει δυστυχώ την καταληκτική ημερομηνία για την κατάθεση τέτοιου αιτήσεων. Εάν όμω το Σώμα συμφωνήσει μαζί σα, μπορούμε να ξεχωρίσουμε την παράγραφο 27. Το θέτω σε ψηφοφορία στο Σώμα. Ποιοι είναι υπέρ η παράγραφο 27 να ψηφιστεί ξεχωριστά. Ποιοι είναι κατά. Απορρίπτεται. Επομένως, Check. Μ' αρέσει αυτό το τμήμα της διαδικασίας, κάθε διαδικασίας. Εμπρός. Ας κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται με 335 ψήφους. του μπλοκ των ε, τροπολογιών από την αρμόδια επιτροπή. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές εγκρίνονται. Με ονομαστική κλίση η τροπολογία 78. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 85. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 86. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές απορρίπτεται. Η τροπολογία 87 έχει αποσυρθεί. Ψηφίζουμε μόνο για την τροπολογία 20. Τροπολογία 20. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 88. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογίες 29 ως 33. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 89. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογίες 39 με 42. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές εγκρίνονται. Ε, τροπολογία 66. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται. Άρα καταπίπτει η τροπολογία 90. Ε, ψηφοφορία στην ε, τροποποιηθήσα πρόταση. Ποιοι είναι υπέρ. Ποιοι είναι κατά. Αποχές εγκρίνεται και με ηλεκτρονική ψηφοφορία η τελική ψήφος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται με 380 ψήφους. Συγχαρητήρια στον κύριο Άλβαρο. Και τώρα έχουμε επεξηγήσεις ψήφου. Στην έκθεση Τράουτμαν η κυρία Ρόιτοβ για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ.